και έχω κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω από πλευράς Συμβουλίου. Έλαβα και την θέση του Συμβουλίου και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τρεις μήνες προθεσμίες από την αυριανή ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου. Έχει τη διάθεση του το Κοινοβούλιο τα πρακτικά του, της συνεδρίας.